χρειάζεται είναι με ενιαία φωνή η οποία θα προκύπτει όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και του θεσμούς αλλά από όλα τα κράτη-μέλη να στηρίξει την τύχη του ανθρώπου. Αυτό ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, η συζήτηση για τον Ai Weiwei έκλεισε. Θα ψηφίσουμε αργότερα σήμερα αφού τελειώσουμε και με τι συζητήσει για τα άλλα δύο κατεπίγοντα θέματα που μας απασχολούν. Το Επόμενο θέμα είναι η απαγόρευση των εκλογών της εξόριστης ε, κυβέρνησης στο Νεπάλ και δίνω τον λόγο στον κύριο Πάσκα για να μας παρουσιάσει το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε την κατάσταση, ξέρουμε πώς έχει και γνωρίζουμε ότι οι Θεβετιανοί προσπαθούν να ορίσουν την τύχη τους. Ο Δαλάη Λάμα είπε ότι θα παρετηθεί και δυστυχώς δεν εξευρέθη μία λύση με τις κινέζικες αρχές. Θεωρούνται λοιπόν ε, ως ε, η μειονότητα αυτή των Θηβετιανών θεωρείται ως πρόσκομα για και κίνδυνος από τις κινέζικες αρχές. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το μεγάλο αυτό, τη μεγάλη αυτή γειτονική χώρα και ε, το Νεπάλ γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι ο βασικός οικονομικός παράγοντας στην περιφέρεια η Το Νεπάλ λοιπόν δέχτηκε αυτές τις πιέσεις και κατέστηλε την εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με την Κίνα που είναι ένας μεγάλος οικονομικός εταίρος. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, με μετά από την καταστολή της απολυταρχίας στο Νεπάλ, στο Κατμαντού, το Νεπάλ και η Κίνα βρίσκονται πολύ πιο κοντά. Άρα οι αρχές του Νεπάλ δεν επέτρεψαν στους θιβετιανούς εξόριστους να ψηφίσουν για την εκλογή ενός νέου πρωθυπουργού. Το ίδιο έγινε και πέρσι τον Οκτώβριο. Οι αστυνομικές αρχές του Νεπάλ δεν επέτρεψαν τις εκλογές μετά από εντολή της Κίνας. Δεν επιτρέπουν δηλαδή σε ένα κυρίαρχο ε, κράτος να δράσει ελεύθερα. Αυτό είναι παρανοϊκό. Η Κίνα έχει τονίσει ότι δεν θα δεχτεί το Δαλάη Λάμα, ο οποίος ζητά αυτονομία και όχι ανεξαρτησία. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή όχι μόνο με τις, ε, κοινωνικές, με τις κινέζικες αρχές αλλά και με τις αρχές του Νεπάλ. Αυτό το νέο καθεστώς μπόρεσε να επιβιώσει εξαιτίας της συνεισφοράς των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Νεπάλ βρίσκεται σε μια ευαίσθητη θέση γεωπολιτικά και κυρίως γεωγραφικά, αλλά θα πρέπει να αντλήσει από το παράδειγμα της Ινδίας και όχι από τον Βορρά, δηλαδή τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική. Ευχαριστούμε, κύριο Τάνο. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάνοκ. Ε, χρησιμοποίησατε 1,5 λεπτό μόνο. Ναι, το ξέρω ότι έχετε δύο. Όταν θα ξανέχετε το λόγο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 37 δευτερόλεπτα. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Δεν φαίνεται να αρκεί η καταστολή των Θιβέτιανων στην Κίνα από τους, ε, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί άρδιν. Δεν επιτελέστηκε καμία πρόοδος, αλλά τώρα φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη καταστολή, οι θηβετιανοί εξόριστοι δεν μπορούν να εκλέξουν ούτε καν την κυβέρνησή τους στην εξορία. Κάτι τέτοιο δεν στάθηκε δυνατόν. Εδώ και πολλά χρόνια είδαμε ότι έχει ασκηθεί μεγάλη πίεση προς τον Νεπάλ μέσω των προσφύγων όταν ανέκυψε ένα τέτοιο ζήτημα, δηλαδή των δικαιωμάτων των Θηβετιανών. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε οι ευρωπαϊκές αρχές να φτάσουν στα σωστά διδάγματα. Οι κινέζικες αρχές καταπιέζουν και το ε, αδελφό κόμμα στο Νεπάλ. Φτάνουν ακόμα και σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Όιλαντ είναι ο επόμενος Ευχαριστώ πολύ. Τρία σημεία θα ήθελα να θέσω για τις ε, τροπολογίες των φιλελευθέρων για το σημείο αυτό. Καταρχήν, η δικαιολόγηση αυτών των τροπολογιών έχει να κάνει με τον αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο έχει ε, ε, προχωρήσει στην κατοχή των, της χώρας του Θιβέτ από την Κίνα. Θα γίνουν λοιπόν όντως εκλογές στο Νεπάλ για θηβετιανή κυβέρνηση. Εντάξει, δεν λαμβάνουμε όμως υπόψη το τι γίνεται με το ίδιο το Θιβέ, το οποίο είναι ακόμα υπό κινέζικη κατοχή. Για ποιο λόγο πιέζουν οι Κινέζοι την κυβέρνηση του Νεπάλ. Μήπως θα μπορούσαμε να μιλάμε πάλι για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς βέβαια να χρειαστεί να αναφερθούμε στη δολοφονία του Αρχιδούκα που τον προκάλεσε. Και τρίτον, το τι σημαίνει η αυτονομία για το Θιβέτ. Νομίζω ότι είναι η μόνη επικοδομητική πρόταση στην οποία θα μπορούσε να υποβάλει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα όπως η αναστολή απαγόρευση των εκλογών ε, στο Νεπάλ για τους Θιβέτ Η κυρία Κέριγκερ Όντεμπερ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Η χώρα από την οποία προέρχομαι έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από ε, κυβερνήσεις στο εξωτερικό. Από το 15 πρόεδροι 15 πρωθυπουργοί και 6 πρόεδροι Πολωνία έχουν ζήσει εξόριστοι και εμείς πάντοτε ζητούσαμε αλληλεγγύη και ζητούσαμε μία λευκή κάρτα για να μπορούμε να ψηφίσουμε όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο μέχρι το 1990 που ξανά γίνεται δημοκρατική η χώρα μας. Αυτή τη στιγμή το Νεπάλ έχει μια ευκαιρία να ξαναξεκινήσει τα όσα κάνει και σύμφωνα με τα όσα λένε στο Σύνταγμα από τις 28 Μαΐου ε, η χώρα θα είναι πλέον μια δημοκρατία. Γιατί λοιπόν να μην επιτρέψει και στις θηγατιανές μειονότητες να ψηφίσουν. Γιατί να χαλάσει τη γιορτή. Μήπως τους βγάζαμε μια κόκκινη κάρτα για να τους πούμε ότι αν δεν αφήσουν τους θηγατιανούς να ψηφίσουν τον ΕΠΑΛ θα κάνει κάτι το παράδεκτο παραβιάζοντας τα βασικά ανθρώπινα, τα θυμολία, ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών ε, στη καταγωγή. καταγωγής. Μήπως θα μπορούσαμε εμεί κάπω να εξουδετερώσουμε την πίεση που ασκεί στον Νεπάλ η Κίνα, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στου Θεβετιανού να συγκεντρώνονται, να εκφράζονται ελεύθερα και να ψηφίζουν. Γιατί στην Πολωνία δεν κατάφεραν να φημώσουν αυτού του πρωθυπουργού και του προέδρου, οι οποίοι κρατούσαν τη φλόγα ζωντανή. Γι' αυτό θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Το Νεπάλ και η Κίνα θα πρέπει να θυμούνται τι έχουμε περάσει εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαν είναι ο επόμενος ομιλητής. Στις 20 Μαρτίου, 8 χιλιάδες ε, Θηβετιανοί έλαβαν μέρος στις ε, εκλογές ε, για την, εξο... στην εξόριστη κυβέρνηση για να ψηφίσουν πρωθυπουργό. Εμείς πήγαμε ως παρατηρητές στις εκλογές αυτές και αυτό που είδαμε και αυτό που παρατηρήσαμε ήταν πως οι εκλογές αυτές έγιναν με ελεύθερο τρόπο και με σεβασμό όλων των δημοκρατικών κριτηρίων. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να γίνουν σεβαστές. Τώρα όμως το Νεπάλ υπό την πίεση των ε, Κινέζων δεν επιτρέπει τη συμμετοχή χιλιάδων Θηβετιανών που ζουν στο Νεπάλ. Παρατείνονται λοιπόν τα μέτρα τα οποία έχουν ε, εμφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πως τα εκλογικά τμήματα τα έκλεισαν και απαγόρευσαν τη διεξαγωγή των εκλογών. Οι Κινέζοι επηρεάζουν βεβαίως το Κατμαντού και θέλουν όλες αυτές οι ελευθερίες του συγκεντρώνεις, τα κτλ. να ε, παραβιαστούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το επιτρέψουμε και θα πρέπει να επιμείνουμε πως θα πρέπει να, γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Μαν. Έχουμε λοιπόν την κυρία Μπασέσκου εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρο. Η απαγόρευση ελευθέρων εκλογών από τις αρχές του Νεπάλ για την ανάδειξη μιας κυβέρνησης στο Νεπάλ των Θιβετιανών εξόριστων είναι κάτι το απαράδεκτο. Έπρεπε να επιτραπούν έτσι ώστε να υπάρχει εκδημοκρατισμός των αρχών. Θα έπρεπε να επιτραπεί αυτή η διενέργεια. Φαίνεται ότι το Νεπάλ δείχνει ότι η δημοκρατία δεν είναι απόλυτη. Βεβαίως ακολουθήθηκε οι δημοκρα... δημοκρατικές εκλογές και θα έπρεπε να επιτρέψει και την διεξαγωγή εκλογών για τους Θηβετιανούς εξόριστους. Θα ήθελα να κάνω έκκληση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή έτσι ώστε να προωθηθεί μια σωστή πολιτική γειτονία σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο εξ στον. των Σαλστών. αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αγωνιστούμε για τα δημοκρατικά δικαιώματα όχι μόνο στη γειτονιά μας, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Πρέπει να έχουμε μια πάγια ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στι μη δημοκρατικά εκλεγμένε κυβερνήσει, απέναντι στι κυβερνήσει που δεν σέβονται τα δημοκρατικά δικαιώματα. Και είπε ο κ. Φερχόφστατ ότι είμαστε υποκριτέ κατά κάποιο τρόπο. Αληθεύει, πάνω από το εμπόριο συχνά δεν βάζουμε καμιά άλλη αρχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η συμφωνία στο Μερκοσούρ, που για χάρη του ανοίγματο του εμπορίου θυσιάζουμε ευχαρίστω το 11% του Αμαζονίου αλλά και εκατομμύρια Ευρωπαίου αγρότε. Σε όλα αυτά φταίει και η Επιτροπή, κύριε Επίτροπε πολλέ φορέ ο επίτροπο εμπορίου δεν αδιαφορεί για τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ πολιτικέ. δεν μπορούμε να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτέ αν συνεχίσουμε έτσι. πρέπει το νεπάλ να σεβαστεί τα δημοκρατικά δικαιώματα των προσφύγων από το θιβέτ πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να χρησιμοποιήσει όποιο μέσο μπορεί να το θέσει αυτό το ζήτημα σε όλα τα πλαίσια και όχι μόνο ε, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. αυτό δεν είναι μόνο θέμα της κυρίας άστον είναι το ίδιο θέμα και του κυρίου de και όλης τη επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρίσμπεκ, μέρος των φιλελευθέρων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζουν την κυβέρνηση του Νεπάλ οι Κινέζοι και για το λόγο αυτό έπεισε τον Νεπάλ να απαγορεύσει τις εκλογές. Αυτό σημαίνει πως στη δίωξη των Θηβετιανών βρήκε νέο σύμμαχο το Κίνα και αυτός ο νέος σύμμαχος είναι το Νεπάλ και όλα αυτά ξεπερνάνε τις εκλογές γιατί εδώ και χρόνια η κυβέρνηση του Νεπάλ υπό την πίεση των κινέζικων αρχών περιορίζει χωρίς τέλος το δικαίωμα έκφρασης των Θηβετιανών που ζουν εξόριστοι στο Νεπάλ και μάλιστα πρόσφυγε του Θιβέτ παραδόθηκαν στους Κινέζους από τον Νεπάλ. Είχαμε συλλήψεις, απαγόρευση διαδηλώσεων, προληπτικές συλλήψεις, απαγόρευση μετακίνησης. Αυτά όλα αποτελούν πολύ συνηθισμένα φαινόμενα για τους Εθιανούς στο Νεπάλ. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε πλέον υποκριτές και να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε αυτές τις πράξεις καταπίεσης του Νεπάλ και τις υπερβολικά πολλές καταπατήσεις της σύμβασης για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να πούμε στο Νεπάλ πως δεν επιτρέπεται πλέον να μεταχειρίζεται άσχημα τους πρόσφυγες, αλλά θα πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματά Είναι πολύ λυπηρό αυτό που διαπιστώνουμε κυρίως για τη χώρα αυτή υποδοχής που είναι το Νεπάλ και που πάντα για τους Θηβετιανούς μέχρι πρόσφατα ήταν ένας τόπος ε, εξορίας. Ο κύριος Ρωμέ Βαϊρουέδα εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ και εγώ πιστεύω πως οι Θεβετιανοί που ζουν στο Κατμαντού δεν έλαβαν δικαίωμα, δεν έλαβαν άδεια να ψηφίσουν στις εκλογές γιατί πίεσε η Κίνα. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο. Η πίεση προς τον Επάλ από την πλευρά της Κίνας που δεν επιτρέπει στους πρόσφυγες να έχουν και να χρησιμοποιούν τα δικαιώματα που θα πρέπει να τους εξασφαλίζει το διεθνέ δίκαιο πρέπει να καταδικαστεί και θα πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας όχι μόνο για τα γεγονότα αυτά αλλά και για το γεγονός πως η, η Κίνα πιέζει, πιέζει τη χώρα του Νεπάλ και δεν τους επιτρέπει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στα άτομα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ε, αντιπροσωπείας στο Κατμαντού θα πρέπει να παρακολουθήσει την κατάσταση και κάτι το οποίο ζητάμε εδώ και πολύ καιρό και καταλαβαίνω πως η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε είναι και ανοίγω εδώ μια παρένθεση, η πίεση της Κίνας είναι κάτι το οποίο πρέπει με όλες μας τις δυνάμεις να αντικρούσουμε και αν δεν το κάνουμε σήμερα όταν ξεκινήσει ο διάλογος μαζί τους φοβάμαι πως δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ακουστούν δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταβάρης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι φοβερό το γεγονός ότι οι Θηβετιανοί δεν έχουν δικαίωμα ε, αυτόβουλης, ε, μάλλον δεν έχουν δικαίωμα αυτοκυριαρχίας στη δική τους χώρα. Δεν έχουν δικαίωμα ούτε στην εξορία από ό,τι φαίνεται, στην οποία έχουν εκδιωχθεί. πολλοί ήταν οι επικριτές των ε, Θιβετιανών. Είπαν ότι ο Δαλάη Λάμα δεν είναι μία δημοκρατικά εκλεγμένη αρχή. Τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει η διαδικασία εκδημοκρατισμού, φαίνεται ότι το Νεπάλ δεν επιτρέπει ούτε καν τη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών, ούτε καν για μία κυβέρνηση εξορίας. Εμείς Είμαστε οι πρώτοι που υποχωρούμε έναντι των Κινέζων μέσα στα πλαίσια οικονομικών καθαρά συμφερόντων. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και τον Νεπάλ ήθελε να κάνει το ίδιο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πιέσουμε τον Νεπάλ θα πρέπει να αρχίσουμε από τα του οίκου μας, δηλαδή να μην δεχόμαστε εμείς τις πιέσεις των ε, Κινέζικων αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ο κύριος Κόβατς. Θα έπρεπε να είναι ο επόμενος ομιλητής, αλλά δεν παρίσταται. Άρα δίνω το λόγο στην κυρία Μακοβέη. Κυρία Μακοβέη, έχετε το λόγο. Η καταστολή των κινέζικων αρχών δεν επέτρεψε τη διενέργεια εκλογών, δεν επέτρεψε σε 82.000 θηβετιανούς εξόριστους να ψηφίσουν το δικαίωμα της ψήφου, το δικαίωμα των ελευθέρων εκλογών είναι ένα βασικό δικαίωμα για κάθε πολίτη και για κάθε κοινότητα. Υπάρχουν πολλά προσκόμματα στη συγκεκριμένη περίπτωση για το να μπορέσει κανείς, για να μπορέσει κανείς να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Είμαι πεπισμένη ότι το Νεπάλ δέχτηκε μεγάλες πιέσεις και οι αρχές του Νεπάλ υπέστησαν μεγάλο εκφοβισμό από τις κινέζικες αρχές. Θα πρέπει εμείς να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη θέση μας και να ασκήσουμε μεγάλη πίεση προς τις αρχές του Νεπάλ και της Κίνας για να δεχτούν το, το, τις δημοκρατικές αυτές εκλογές, τη διενέργειά τους. Βρισκόμαστε στο κάτσε, η κυρία Μισάια ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η πίεση η οποία ασκεί η Κίνα στην κατάσταση στο Νεπάλ έχει φτάσει σε οριακή κατάσταση. Οι Θηβετιανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν καν για 6 στον Πρωθυπουργό και βρίσκονται σε εξορία. Έχουμε λοιπόν πίεση από την Κίνα και πίεση για την πολιτική της μία Κίνας. Για τον λόγο αυτό οι πρόσφυγε από το Θιβέτ βρίσκονται υπό πολύ σκληρό έλεγχο στο Νεπάλ και το ψήφισμα μιλά για την κατάσταση με τις εκλογές, αλλά εδώ προκύπτει και άλλο θέμα ότι δηλαδή η Κίνα έχει καταλάβει τη χώρα τους και τους και τώρα και στην εξορία. Χρειάζεται λοιπόν και εμείς να μιλήσουμε με μία φωνή όταν μιλάμε με την Κίνα. Ο κύριος Κέλλη θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι επρόκειτο να λάβω το λόγο, αλλά επειδή ο Δαλάη Λάμα αυτή τη στιγμή επισκέπτεται τη χώρα μου την επόμενη Πέμπτη και θα μιλήσει στη δική μου εκλογική ε, περιφέρεια στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ, σίγουρα θα πει πολλά και για το θέμα αυτό και για άλλα και η μεταχείριση που έτυχαν ε, οι Θεβετιανοί από την κυβέρνηση του Νεπάλ με την κατάσχεση των εκλογικών ε, καλπών είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα λυπηρό. 10.000 ψήφοι περίπου δεν μετρήθηκαν γιατί εξαφανίστηκαν οι κάλπες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει ομόφωνα να καταδικάσει τα επεισόδια αυτά για να πιέσει όχι μόνο τον ΕΠΑΛ αλλά και τα αφεντικά τους, τους Κινέζους. Έτσι ώστε να δείξουν λίγο μεγαλύτερη κατανόηση και κυρίω για το θέμα του Θιβέτ και του Δαλάη Λάμα. Και θέλω να χαιρετήσω την παρουσία του στην Ιρλανδία. Θα έρθουν επίσης και η Βασίλισσα της Αγγλίας και ο Πρόεδρος Ομπάμα. Ο κύριος Ρέπο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το δικαίωμα να μιλήσω και εξίσου σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να, να... Με συγχωρείτε, να ψηφίσει ελεύθερα για να μπορεί κανείς να διατηρήσει λοιπόν την ε, πολιτιστική του ταυτότητα. Οι Θιβετιανοί έχουν επιλέξει την ηγεσία τους. Και νομίζω ότι αν ανατρέξουμε στο 2009 και στη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είχαμε υποβάλει μια δήλωση ζητώντας να στηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να φανούμε συνεκτικοί με τα όσα είχαμε πει τότε και να στηρίξουμε τις πολιτικές μας. Προφανώς το, Θιβέτα, το, το Νεπάλ, με συγχωρείτε, υποκύπτει στις πιέσεις της Κίνας και θα πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι έχουν υπογράψει την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα πρέπει τα δικαιώματα αυτά να τα προσφέρουν στους Ιδετιανούς πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς. Περιμένει να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 20.000 Θεβετιανοί στο Νεπάλ και μπορούν να ασκήσουν με ελευθερία, οικονομική δραστηριότητα και έχουν και κάποια πολιτική δυνατότητα και ελευθερία. Στις 20 Μαρτίου οι εκλογές ήταν πολύ σημαντικές για όλη την κοινότητα των Θηβετιανών που ζουν εκτός του Θιβέτ. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες όσον αφορά τις πολιτικές δυνάμεις και την κυβέρνηση στο Νεπάλ που περιορίζουν την δραστηριότητα των Θηβετιανών. Αυτό δεν έγινε για πρώτη φορά και σε άλλες εκλογές στις 3 Οκτωβρίου του 2010 υπήρξε περιορισμός όσον αφορά τα εκλογικά δικαιώματα των Θηβετιανών που ζουν στο Νεπάλ. Και ξέρουμε ότι αυτό βεβαίως γίνεται από κοινού με την κυβέρνηση του Νεπάλ. Ξέρουμε επίσης ότι ο περιορισμός της ελευθερίας ε, των μελών της κοινότητας ε, του Τιβέτ, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τύχουν τις προσοχή μας και η δυνατότητα να έχει κανείς ελεύθερη πρόσβαση στο Νεπάλ θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να προστατευθούν οι πρόσφυγες, οι Θεβετιανοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους προς το Κατμαντού θα πρέπει να προστατευθούν και να μπορέσουν να φτάσουν εκεί χωρίς ε, εμπόδια και δυσκολίες και να μπορέσουν να καταχωρηθούν ε, στα μητρώα των ε, κατοίκων του Νεπάλ. Εμείς βεβαίως και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα προετοιμάσουμε νέα έκθεση στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τέλος της συζήτησης και βεβαίως θα ψηφίσουμε ακριβώς μετά το τέλος του τελευταίου κατεπήγοντος θέματος που είναι η κατάσταση στην Ζιμπάμπο.